Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σε συνεδρίαση της 12 η Ιουλίου προέβη στον έλεγχο της εντολής του κυρίου Τζον Φλακ και πρότεινε ομόφωνα να εγκριθεί η εντολή αυτή από τις 28 Ιουνίου 2017. Επίσης, συνεδρίαση της 7, 7 Σεπτεμβρίου 2017 η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της εντολής των Έλισεν, Λεσεβαλιέ, Βιού Καν και Όαρθ